ich eröffne die sitzung des haushaltskontrollausschusses. ich begrüße sie sehr herzlich. guten morgen in straßburg. Καλημέρα σας. Ξεκινούμε τη συνεδρίασή μας εδώ στο Στρασβούργο. Καλωσορίζουμε τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και πρώην συνάδελφο Αλεξάνδερ Στούπς. Χαίρομαι, χαίρομαι ιδιαίτερος που είστε εδώ. Έχετε την ημερήσια διάταξη, αλλαγές δεν προβλέπονται. Έχετε από το News ε, τα στοιχεία και για τη διερμηνία βεβαίως και το γεγονός ότι μεταδίδεται μέσω του διαδικτύου η συνεδρίασή μας όπως πάντα. Η κυρία Μογκερίνη νοσεί δυστυχώς. 25 Ιανουαρίου, την προσεχή δηλαδή Πέμπτη, θα έρθει για να μας συναντήσει. Στις 9 το πρωί ξεκινάει η συνεδρίαση και γι' αυτό και διατηρείται αυτή η συνεδρίαση. Και βεβαίως ευχόμαστε ταχύτατη ανάρρωση στην κυρία Μογκερίνη. Έτσι λοιπόν έχουμε την έκθεση, τη έκθεση 2016 της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Ε, και έχουμε το θέμα των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, της ε, βιώσιμης ανάπτυξης, διαφάνεια, ένα πληρέστατο φάκελο τεκμηρίωσης που μα διαβιβάζει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων για και είναι πολύ σημαντικέ πληροφορίε Για την ετήσια έκθεση έχουμε τον κύριο Βάλλη Αρμόδιο. Δίνω το λόγο πρώτα στον κύριο Στούμπα και σας ευχαριστούμε που είστε εδώ. Σα ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε και ευχαριστώ για τα ευγενικά σας λόγια. Χαίρομαι πολύ που ξαναβρίσκομαι εδώ γιατί διτέλεσα και Ευρωβουλευτής και μέλος Επιτροπής Ελέγχου Προϋπολογισμού από το 2004 μέχρι το 2008. Και θυμάμαι αν τότε είχα ασχοληθεί και με την απαλλαγή για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, αλλά μου διαφεύγει, δεν ξέρω αν εσείς το θυμάστε. Αλλά χαίρομαι που ξανά ήρθα και αν θυμάμαι καλά, ε, έγινα και στα μέσα της θητείας συντονιστής ε, του ΕΛΚ όταν ε, ασχολούμαστε με τα θέματα αυτά. Και θεώρησα συναρπαστική τη συμμετοχή μου στην Επιτροπή Ελέγχου Προπολογισμού και, και μάλιστα 8 χρόνια ήμουν στην κυβέρνηση ω Υπουργό Εξωτερικών, Υπουργό Οικονομικών και Πρωθυπουργό. Έχω 8 χρόνια πείρα κυβερνητική και ελπίζω να αντιλαμβάνεστε πόσο ε, σε πόση σε την προνομιακή θέση είστε ως Ευρωβουλευτές, γιατί το έργο σας είναι εξαιρετικά σημαντικό και η η επιρροή που έχουμε σε σχέση με εθνικού ευρωβουλευτέ, ακόμη και σε σχέση με υπουργού, ε, η δική σας επιρροή είναι τεράστια. Και πολύ αργό γίνεται σε νομοθετικέ επιτροπέ. Αλλά όπω ξέρουμε, επιτροπέ ε, προπολογισμών και ελέγχου προπολογισμού ίσω είναι από τι πιο σημαντικέ ε, επιτροπέ του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χαίρομαι πραγματικά ειλικρινά που ξαναβρίσκομαι εδώ και νιώθω σαν στο σπίτι μου. Πολύ ενδιαφέρουσα αυτή η μέρα για αυτή τη συζήτηση. Γιατί όσο εμείς μιλάμε, ο πρόεδρος Βέρνερ Χόιερ θα παρουσιάσει τα αποτελέσματα της ΕΤΕ για το 2017. Και στη συνέχεια στις ε, ερωταπαντήσεις, ε, πολύ ευχαρίστω να σας δώσω κάποια σχετικά στοιχεία από τα αποτελέσματά μας για το 2017. Πριν ε, περάσω στην ομιλία μου και θα ήθελα να πω ότι επειδή ασχολούμαι μανιωδώς με την Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι η ΕΤΕ είναι το πιο καλά κρατημένο μυστικό της Ευρωπαϊκής Ένωσης και πραγματικός φιλοευρωπαίος και ως υπέρμαχος ε, του έργου της Ευρωπαϊκής Ένωσης είτε για το κλίμα, το περιβάλλον, για τις υποδομές, για την καινοτομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις πιστεύω ε, ό,τι και να πούμε προωθεί ουσιαστικά το έργο της ΕΤΕ. Λίγοι γνωρίζουν ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είναι η μεγαλύτερη πολυμερής τράπεζα του κόσμου. Είναι τριπλάσια από την Παγκόσμια Τράπεζα και δεκαπλάσια από την Τράπεζα Ενοικοδόμησης και Ανάπτυξης. Και ε, έχουμε 600 δισεκατομμύρια ε, περιουσιακά στοιχεία, στοιχεία του ενεργητικού. Τα δικά μας, τις εννοώ τα δικά σας, 600 δις. Το κεφάλαιο μας είναι 250 δισεκατομμύρια ευρώ και δίνουμε ε, δάνεια ύψους 8 δισεκατομμύριων ευρώ, 80 δισεκατομμυρίων ευρώ το χρόνο και με μόχλευση διπλάσια-τριπλάσια φτάνουμε στα 220-250 δισεκατομμύρια ενώ 150 δις είναι περίπου το χρόνο ο κοινοτικό προπολογισμό. Βλέπετε ποιο είναι το τεράστιο δυναμικό της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και αυτό πολύ συχνά το ξεχνούμε. Γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό εσείς να μας ελέγχετε και να μεριμνάτε ότι είναι σωστή η συμπεριφορά μας. Ε, θα σταθώ σε τρία σημεία στην ομιλία μου. Το πρώτο θα είναι τα αποτελέσματά μας για το 2016, το δεύτερο για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το τρίτο για τη διαφάνεια. Θα προσπαθήσω να μην ξεπεράσω το δεκάλεπτο που μου δώσατε. Σε ό,τι αφορά τα αποτελέσματά μας για το 2016, ξέρετε ότι στόχος μας είναι να στηρίζουμε την οικονομία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πολιτικές της και την εσωτερική αγορά. Και θα έλεγα ότι από και η σιανή άποψη τα πήγαμε αρκετά καλά και κατά τη διάρκεια της χρηματοπιστωτικής κρίσης. Και αυτό έγινε χάρη όχι μόνο στην Επιτροπή και το σχέδιο Juncker, αλλά και χάρη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο που ενέκρινε το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ. Και αν δείτε τώρα την ευρωπαϊκή οικονομία, αμέσως μετά που ε, κατέληψε εγώ την κυβέρνηση, πήγε πολύ καλύτερα. Οι οικονομικοί μας δείκτες είναι σχετικά θετικοί, αλλά φυσικά υπάρχει δρόμος ε, και περιθώριο για βελτίωση και θα έλεγα και καινοτομία. Και γι' αυτό έχουμε και την ΕΤΕ. Και αν δούμε τα, τα αποτελέσματα για το 2006 για την καινοτομία, το 2016 δώσαμε χρηματοδομικά μέσα εγγυήσεις σε δάνεια 83 83,8 δισεκατομμύρια ευρώ. 83,8 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, και μάλιστα σε τέσσερις κατηγορίες μοιράστηκαν αυτά. Περιβάλλον και κλίμα, περίπου 17 δισεκατομμύρια. Υποδομές, περίπου 20 δισεκατομμύρια για την καινοτομία 13,5 δισεκατομμύρια ευρώ και για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις περίπου 34 δισεκατομμύρια δώσαμε σε χρηματοδοτικά μέσα, δάνεια, και και ούτω καθεξής. Ε, έτσι φτάνουμε περίπου στα 83,8-84 σχεδόν δισεκατομμύρια. Και αν σε αυτό προσθέσουμε τη μόχλευση, ε, καταλήγουμε σε πολύ υψηλότερα ποσά, περίπου στα 280 δισεκατομμύρια ευρώ, ε, προσπαθώντας να γεφυρώσουμε κάποια κενά της αγοράς. Ε, οπότε, ουσιαστικά έχουμε 790, 787 ουσιαστικά ε, ενέργειες, επιχειρήσεις ή δάνεια. Με, μερικοί μας είπαν τα κόκκινα σας δάνεια τι ύψος έχουν, 26 είναι και 0,4% της συνολικής αξίας για τα κόκκινα, τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια. Έχουν χαμηλότερο το ποσοστό μη εξυπηρετούμενων δανείων, μπορώ να σας πω το χαμηλότερο ποσοστό οποιασδήποτε τράπεζα του κόσμου. Οπότε και με αυτή την άποψη των μη εξυπηρετούμενων δανείων ήμασταν πολύ τυχεροί. Έγινε μάλιστα και μια μελέτη επιπτώσεων εξωτερική για τα, έτη 2016 και 2017 και τα στοιχεία που μας δίνει η μελέτη αντικτύπου είναι τα εξή. Με βάση τη σχετική εξωτερική μελέτη, το έργο και οι επενδύσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων έδωσαν 2,27 δισεκατομμύρια νέες θέσεις εργασίας και επιπλέον 2,3% αύξηση του ΑΕΠ στην ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Βέβαια, μπορεί κανεί να αμφισβητήσει τα οικονομετρικά στοιχεία αυτών των αριθμών. Αλλά το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων συμμετέχει σε κάποια σχέδια, προσέλκυσε επενδύσεις και δημιουργήσαμε έτσι 2,25 εκατομμύρια θέσεις απασχόλησης και αυξήσαμε 2,23% του ΑΕΠ μέχρι το 2020. Τώρα για το 2017 περίπου παρόμοια στοιχεία έχουμε και θα τα αναπτύξω δεχομένως στην ακόλουθη συζήτηση. Λίγα λόγια για το ΕΦΣΥ, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Εγώ θεωρώ ότι το ΕΦΣΥ είναι από τους καλύτερους νεοτερισμούς της Ευρωπαϊκής Ένωσης εδώ και πολλά χρόνια. Η δική μου άποψη είναι και όλοι παρακολουθείτε τον υπολογισμό, όλοι είστε Ευρωπαίοι. Εγώ θεωρώ ότι το μέγεθος του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού έχει μείνει σχετικά σταθερό Μιλούμε για ένα περίπου τα εκατό του ακαθάριστου ε, ε, εθνικού εισοδήματο πάνω κάτω και θα έχουμε και τις συνέπειες του Brexit. Το, οπότε αν δεν αυξάνεται το συνολικό ποσό των δανείων και των επιχορηγήσεων και θέλουμε κάποια προστιθέμενη αξία, τι κάνουμε, ε, προσθέτουμε κάποια χρηματοδοτικά μέσα και κάποιες δημοσιονομικές εγγύσεις. Αυτό έκανε το ΕΦΣΥ και ήταν πολύ θετική η συμμετοχή και η συνεισφορά του ΕΦΣΥ και μάλιστα ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στα θέματα αυτά ήταν ε, πολύ σημαντικός. Όλοι γνωρίζετε το ΕΦΣΥ. Από τα μέσα του 2018 θα δημιουργήσει, θα, θα παράγει 350 δισεκατομμύρια ευρώ και 500 δισεκατομμύρια μέχρι το 2020. Και μάλιστα ακολουθούμε τους, την πορεία και θα υλοποιήσουμε τους στόχους. Τα πρώτα στοιχεία από τα μέσα Σεπτεμβρίου μας δείχνουν ότι τον Σεπτέμβριο του 2017 είχαμε 256 δισεκατομμύρια που έχουν παραχθεί ουσιαστικά από το ΕΦΣΥ και έχουμε υλοποιήσει μέχρι στιγμής το 82% του στόχου. Ε, μέχρι τα τέλη του καλοκαιριού θα έχουμε υλοποιήσει το έπακρο το στόχο. Και από αυτή την άποψη το ΕΦΣΥ στέφθηκε με επιτυχία. Επίσης, το ΕΦΣΙ καθιστά την ΕΤΕ πολύ πιο ρηψοκίνδυνη γιατί παλιά υιοθετούσαμε μόνο 450 ε, μεγαλεπίβολα μακρόπνοα σχέδια ασφαλή. Τώρα έχουμε πολύ περισσότερα και μερικά είναι και πολύ πιο ρηψοκίνδυνα από ό,τι στο παρελθόν. Οπότε εντό τη Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων είχαμε ανέκαθεν κάποια διστακτικότητα, επιφυλακτικότητα απέναντι στο ρίσκο, τον κίνδυνο. Τώρα χάρη στην υποστήριξη και το ΕΦΣΥ μπορούμε να αναλαμβάνουμε και πιο τέτοια επικίνδυνα σχέδια. Έχουμε και συνεργασία με τις Εθνικές Τράπεζες Προώθησης. Έχουμε 25 μνημόνια συνεννόησης με Εθνικές Τράπεζες Προώθησης, κάτι που μας έφερε πιο κοντά στις τράπεζες αυτές. Και αν θα μπορούσα να προδικάσω, να προεξοφλήσω κάποιες ε, απορίες σας, για παράδειγμα για την κατανομή των κονδύλιων και ποιοι είναι οι δικαιούχοι. Να σας δώσω συγκεκριμένα στοιχεία και γι' αυτό, αλλά πρώτα θα ήθελα να τονίσω ότι δεν έχουμε ποσοστώσεις, ούτε στο ΕΦΣΙ ούτε πουθενά άλλου. Δεν δίνουμε κονδύλια σε συγκεκριμένες χώρες. Όσο φυσικά μεγαλύτερη είναι χώρα, τόσο μεγαλύτερος είναι και ο όγκος των επενδύσεων. Αλλά αν το δείτε σε σχέση με το ΑΕΠ, εκεί είναι πολύ διαφορετικά τα στοιχεία. Η Εστονία, η Πορτογαλία, η Ελλάδα, η Ισπανία, η Λετωνία ε, έχουν τα πρωτεία και υπάρχουν μεγάλες διαφορές. Προσπαθούμε να έχουμε μια ακριβοδίκαιη κατανομή, αλλά ε, το ζητούμενο είναι τα σχέδια. Δεν είναι ότι χρειάζεται περισσότερα χρήματα η Σουηδία ή η Γερμανία. Εξαρτάται από τα σχέδια. Αν ένα σχέδιο δεν έχει προστιθέμενη αξία, αν δεν πληρεί τι ε, προποθέσει τη προσθετικότητα και άλλα κριτήρια, τότε δεν επιλέγεται. Ο αντίκτυπος του ΕΦΣΙ για το 2015 και το 2016, η ίδια εξωτερική μελέτη δείχνει 0,7% του ΑΕΠ και 690.000 θέσεις απασχόλησης, 0,7% του ΑΕΠ και 690.000 νέες θέσει απασχόλησης χάρη στα προγράμματα αυτά. Οπότε το ΕΦΣΙ έχει αποδείξει την αξία του και τη σκοπιμότητά του. Και το τρίτο και τελευταίο σημείο αφορά τη διαφάνεια και τη διακυβέρνηση. Θα λέγαμε ότι βρισκόμαστε στην πρωτοκαθεδρία ε, σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια σε σχέση με άλλα διεθνή χρηματοδοτικά Ινστιτούτα και φορείς. Έχουμε ε, με ένα διοντολογικό κώδικα που ακολουθούμε και τις βέλτιστες πρακτικές. Για το 2016 προσπαθούμε να έχουμε περισσότερες εκθέσεις πιο φιλικές προς το χρήστη, προς τον αναγνώστη. Ευθυγραμμίζουμε τις ενέργειές μας με την ομολογία και την ε, ευρωπαϊκή νομοθεσία. Ε, μας προβληματίζει και το θέμα της πάταξης των απατών, συνεργασία με την Όλαφ. Φυσικά αντιλαμβανόμαστε το εύλογο αίτημα για αυξημένη διαφάνεια και χαιρόμαστε που η Επιτροπή σας μας ζήτησε να δημοσιεύουμε τις συνεδριάσεις, τα πρακτικά των συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου και το κάναμε. Προσπαθούμε να είμαστε όσο πιο διαφανείς γίνεται, προσπαθούμε να βελτιώσουμε την επικοινωνιακή μας πολιτική και την επικοινωνία μας, αλλά υπάρχουν και κάποιες υποθέσεις ιδιαίτερα επενδύσεων που δεν μπορούμε να είμαστε τόσο διαφανείς όσο θα θέλαμε. Αλλά αυτή είναι μια ισορροπία που προσπαθούμε να κρατούμε ανα πάσα στιγμή. Οπότε έρχομαι στα τελικά μου σχόλια. Το 2016 ήταν μια καλή χρονιά για μας, ε, θετική χρονιά για την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, παρά τον Brexit, παρά τον Τραμπ. Από τραπεζική άποψη ήταν καλή χρονιά το 2016. Οι δείκτες και τα στοιχεία είναι καλά, τους στόχους μας τους πραγματοποιήσαμε Τώρα, αν με ρωτήσετε για το 2017, να σας δώσω κάποια στοιχεία. Και πέρυσι είχαμε καλή χρονιά στην ΕΤΕ. Εγώ θεωρώ προσωπικά ότι έχουμε τρεις μείζονες προκλήσεις για το 2018. Η παριθμόν ένα πρόκληση είναι το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο μετά το 2020 και πολύ ευχαρίστω να αναπτύξω και αυτό μετά στη συζήτηση. Το δεύτερο είναι η συζήτηση που εξελίσσεται για ένα παράρτημα της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων ε, της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Ανάπτυξης εντός της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και ε, τα, η επιχειρησιακή μας στόχη είναι το τρίτο σημείο. Κάτι που ανέκαθεν προσπαθούμε να τηρούμε και να υλοποιούμε. Αυτά ως προς τα αποτελέσματα του 2016, το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων και το τρίτο θέμα, την διαφάνεια και τη διακυβέρνηση. Ευχαριστώ. Ναι, ευχαριστώ πολύ και εγώ και εμείς χαιρόμαστε σου. Και θυμάμαι όντως ε, τις εποχές εκείνες που ήσουν στην Επιτροπή Ελέγχου του προϋπολογισμού. Μια ωραία εποχή. Και έτσι μπορέσαμε να στήσουμε κιόλας αυτή τη δουλειά. Ο Σανφος Βάλης, ηγητής, έχει το λόγο. Ναι, ευχαριστώ Πρόεδρε. Και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Στουπ που είναι εδώ και για την έκθεσή του βεβαίω. Ιδιαίτερα ευχαριστώ για όλα τα στοιχεία που μου προσφέρατε και από τις πρώτες μου επαφές με την ε, Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων ε, για τα μέχρι τώρα αποτελέσματα στον έλεγχο του προϋπολογισμού και που βέβαια θα ενσωματωθούν ε, και στην έκθεση και πιστεύω ότι και οι συνάδελφοι συμμερίζονται αυτή την προσέγγιση. Άπαξ και υπάρχει ένα ζήτημα δηλαδή να προσπαθούμε με την ΕΤΕΠ να το συζητούμε και να προχωρήσουμε στην εξέταση και μετώπιση των πραγματικών ε, προβλημάτων σε σχέση με το έτσε τη ζήτημα και γεωγραφικής ε, ένδειξης που θα πρέπει ενδεχομένως χάρη σε στατιστικά στοιχεία, σε καλύτερα στατιστικά στοιχεία που θα αναφέρονται και στο ΑΕΠ, ε, την κατανομή του πληθυσμού, τη γεωγραφική κατανομή στις διάφορες χώρες να μεταστραφεί σε μια προσέγγιση που δεν θα έχει μόνο ποσοτικό χαρακτήρα και δεν θα αφορά μόνο χρηματικά ποσά. Για την έκθεση αυτή, λοιπόν, την ετήσια έκθεση 2016, θέλω να υπενθυμίσω στην ΕΤΕΠ ότι χρήσιμο θα ήταν και απαραίτητο να λεβληθούν υπόψη και να λαμβάνονται πάντα υπόψη οι παρατηρήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Χρειάζεται μια μεγαλύτερη προσπάθεια προ την κατεύθυνση αυτή. Ακριβώ σε ε, θέμα ε, έκθεσης της ΕΤΕΠ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο έχει εγερθεί το ζήτημα της ε, κάλυψης όλων των τύπων πληροφοριών γιατί βλέπουμε ότι είτε πρόκειται για στατιστική είτε για δημοσιονομική λειτουργική έκθεση ε, τίθεται για εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ε, έχουμε μεγάλη πληθώρα στοιχείων και καλό θα ήταν όλα αυτά να ενωθούν σε ένα έγγραφο για να είναι πιο ευανάγνωστα. Και επίσης ε, η ΕΤΕΠ όχι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση αλλά και σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες διαδραματίζει πρωταγωνιστικό ρόλο με 25% των επενδύσεών της ε, στην ε, στόχευση της βελτίωσης αποτελεσματικότητας στη χρήση ενέργειας και σε αυτό θα πρέπει να συνεχιστούν οι προσπάθειες. Θα πρέπει, πιστεύω, να καταγραφεί πιο αποτελεσματικά η δουλειά που κάνει η ΕΤΕΠ σε σχέση με το Ταμείο ΕΤΣΕ. Για τα στοιχεία που μας δίνει η ΕΤΣΕ μας δείχνει ένα ε, μάλλον θα έπρεπε να έχουμε ένα 25% και ακόμη μεγαλύτερο τμήμα ε, απόδοσης επένδυσης, αλλά είμαστε σε ποσοστά χαμηλότερα με βάση τα στοιχεία που μας έχουν χορηγηθεί. Πρέπει λοιπόν τα διαθέσιμα χάρη στο έτσι κονδύλια ε, να ενισχυθούν, να μόχλευθούν και ιδιαιτέρως ε, στο θέμα της ε, ενέργειας πρέπει να προχωρήσουμε σε αποτελεσματικότερη χρήση της και σε εγκατάλειψη των ορυκτών καυσίμων. Ιδάλλως θα χρειαστεί όλοι μας να μεταναστεύσουμε κάποια στιγμή σε άλλο πλανήτη. Αυτό που κάνει η ΕΤΕΠ λοιπόν πρέπει να συνεχίσει να το κάνει χωρίς να δέχεται ε, ή να υφίσταται πιέσεις από κυβερνήσεις ή μεγάλα μεγάλους διεθνείς οργανισμούς ή και διεθνείς ε, πολυεθνικές επιχειρήσεις που επιμένουν σε επενδύσεις που δεν έχουν αποδοτικότητα. Σε σχέση με τη δημοσιονομική πολιτική και τη διαφάνεια, πολύ σημαντικό και για το Κοινοβούλιο το θέμα αυτό, η ΕΤΕΠ θα πρέπει να υιοθετήσει περαιτέρω διατάξεις που θα ενισχύσουν τη διαφάνεια, τη φορολογική, να μην ε, επιτρέπει την δράση κάποιων παραγόντων που προσπαθούν να αποκρύψουν στοιχεία ή που έχουν συνάφεια με φορολογικούς παραδείσους. Είναι πολύ σημαντικό αυτό για το Κοινοβούλιο να υπάρχουν λογαριασμοί ανακράτος και να ε, τηρούνται απαρέγκλητα όλα τα πρότυπα που έχει οθετήσει και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο στη τελευταία ανάλυση και αυτό βέβαια δεν θα λείψει από την ετήσια μας έκθεση για τον έλεγχο του προϋπολογισμού. Στην έκθεση επίσης είναι θεμελιώδη σημασία να επισημαίνεται η αιρεσιμότητα, η όρη βάση των οποίων θα διατεθούν τα στοιχεία του και η συμπληρωματικότητα, η προσθετικότητα του Ταμείου ΕΤΣΕ, του σχεδίου Juncker. γιατί αυτό είχε ενσωματωθεί στο πρώτο, στην πρώτη έκθεση, ωστόσο με τη δεύτερη ε, προσθέθηκαν και άλλα ε, άλλες απαιτήσει του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου με έμφαση ιδιαίτερα στη διαφάνεια και την προσθετικότητα για το σχέδιο Juncker. Σε αυτά λοιπόν πρέπει να σταθούμε. Και εμείς ως Κοινοβούλιο σας καλούμε να προχωρήσετε στην εφαρμογή του νέου αυτού κανονισμού που πρόσφατα εγκρίθηκε και που απαιτεί συμπληρωματικές και περισσότερες πληροφορίες για το θέμα ιδιαίτερα της προσθετικότητας, γιατί δεν της προσθετικότητας στο σχέδιο Juncker. Ιδάλλως ο κόσμος θα καταλήξει να πιστεύει ότι τη δουλειά αυτή που προσφέρει το έτσι, τις ευκαιρίες που προσφέρει το έτσι, θα μπορούσε ούτως ή άλλως να τις έχει επιτελέσει η ΕΤΕΠ χωρίς το ε, σχέδιο Juncker. Γι' αυτό θα ήταν ε, καλό και μάλιστα ένα πρώτο βήμα θα ήταν να προχωρήσετε σε μια ανάλυση της προσθετικότητας σε σχέση με την ενεργειακή μετάβαση ε, σχέδια δηλαδή και έργα που έχουν χρηματοδοτηθεί σε συνέργεια μεταξύ Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων και άλλων ταμείων. Και ολοκληρώνοντας, θέλω να αναφερθώ στην τεχνική υποστήριξη το 2016 ενίσχυσε τη εργασία στο πεδίο αυτό η ΕΤΕΠ από ό,τι σημειώνω για το χώρο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Θα ήθελα όμω αντίστοιχα και συστηματικά να συμβαίνει το ίδιο και εντό Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί διαθέτει η ΕΤΕΠ και τι δομέ και τι ικανότητε να αναπτύξει ένα δίκτυο ε, παροχής αυτών των υπηρεσιών σε όλη την Ευρωπαϊκή Ένωση στα κράτη-μέλη που έχουν ανάγκη και καλό και τους συναδέλφους να βοηθήσουν στο βαθμό που μπορούν την ΕΒΤΕΠ στην ανάπτυξη αυτού του έργου ώστε να είναι διαθέσιμα τα ε, κονδύλια για τις επενδύσεις παντού. Και αυτό με ιδιαίτερη έμφαση και στη, στο ρόλο που διαδραματίζουν ε, οι, ευρωπαϊκοί, οι εθνικές τράπεζες που προωθούν τις επενδύσεις, όπως σε παραδείγμα στην Ιταλία που έχει πάρα πολύ σημαντικό ρόλο η αντίστοιχη η Promotional National Bank και νομίζω ότι μπορούμε να ε, περιμένουμε περισσότερες επενδύσεις από την ΕΤΕΠ στο πεδίο αυτό. Ουσιαστικά δηλαδή να οθείται η κάθε εθνική κυβέρνηση σε μια μεταρρύθμιση του συστήματος των ιδιωτικών επενδύσεων που διαθέτει σε εθνικό επίπεδο έτσι ώστε να αξιοποιεί όλα τα κονδύλια που διαθέτει η Ευρωπαϊκή Ένωση για την εν λόγω χώρα. Έχω πει πολλά. Για να ολοκληρώσω πρέπει οπωσδήποτε το Κοινοβούλιο να επιληφθεί αυτής της έκθεσης και θέλω να ακούσω τους συναδέλφους πάνω απ' όλα τι γνώμη έχουν για να μπορέσουμε στη συνέχεια να προχωρήσουμε σε μια δημόσια ανταλλαγή απόψεων, γιατί ακόμα την έκθεση του Κοινοβουλίου για το 2016 δεν την έχουμε συζητήσει και θα πραγματοποιηθεί αυτός ο διάλογος στις επόμενες ημέρες. Ευχαριστώ πολύ. Θα δώσω το λόγο στον συνάδελφο Στούμπ, στον κύριο Στούμπ για να απαντήσει. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, ευχαριστώ και τον ε, εισηγητή, τον κύριο Βάλη. Είχαμε εξαιρετική συνεργασία Είχαμε μια σειρά συναντήσεων και μπορέσαμε να ανταλλάξουμε απόψεις μέχρι και χτες. Για τα συγκεκριμένα σημεία που θίξατε, η γεωγραφική κατανομή ήταν η πρώτη σας παρατήρηση. Εννοείται ότι η τράπεζα προσπαθεί να, να είναι όσο πιο αποτελεσματική μπορεί και λαμβάνουμε υπόψη μας τα σχέδια που υποβάλλονται, λαμβάνουμε υπόψη μας την αιρεσιμότητα, ότι ισχύει δηλαδή στις διάφορες περιοχές και την ίδια ώρα πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη μας ε, και την απόδοση των συγκεκριμένων ε, σχεδίων και προγραμμάτων. Βεβαίως πρόκειται για μια τράπεζα μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα, να το πω έτσι. Και πολλές φορές ε, ακούω επιχειρήματα ότι παραδείγματο χάρη φέτο δίνονται περισσότερα ποσά στην Ιταλία, Ισπανία, Γαλλία ή Γερμανία. Αυτό οφείλεται στο μέγεθος των κρατών. Για το Ηνωμένο Βασίλειο ήταν πολύ χαμηλά τα ποσά, τουλάχιστον για το 2017, για ευνόητους λόγους. Απ' την άλλη πλευρά, το ανακεφαλήν ποσό που επενδύεται και ο λόγος, η αναλογία μεταξύ ποσών που δίνονται για επένδυση και του ΑΕΠ και μάλιστα για το 2017. Αν κοιτάξετε τα στοιχεία που έδωσε ο Βέρνερ Χόιερ για το τέλος του 2016 θα διαπιστώσετε ότι τηρούνται ε, πολύ συγκεκριμένες ε, αναλογίες. Όσον αφορά την αποτελεσματικότητα, αναφερθήκατε βεβαίως στο Τραμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Είμαστε νομίζω μία από τις λίγες τράπεζες στον κόσμο που φυσικά και στοχεύουμε να τηρήσουμε τους στόχους για τη βιωσιμότητα, τους στόχους που αφορούν την κλιματική αλλαγή και φυσικά γνωρίζετε και το σχέδιό μας για τα green bonds. Χρησιμοποιούμε λοιπόν κάθε φορά και αυτές τις παραμέτρους όταν ελέγχουμε και εκτιμούμε και αξιολογούμε μια επένδυση. Και σαν υπουργό ε, Οικονομικών πολύ ευαίσθητο αυτό η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βεβαίως και συμμορφώνεται στα λεγόμενα στα λεγόμενα όπκο και φυσικά λαμβάνουμε υπόψη μας και άλλες παραμέτρους όπως θέματα ε, δικαιοσύνης, δίκαιης φορολόγησης, το θέμα της, ε, του BEPS, ε δηλαδή το να υπάρχει έλεγχος του πώς φορολογούνται τα κεφάλαια. Αυτό που είναι πάρα πολύ σημαντικό επίσης είναι το θέμα της προσθετικότητας που θίξατε. Βεβαίως και προσπαθούμε επειδή ακριβώς ε, η αξιολόγησή μας είναι 3α από τους οίκους αξιολόγησης, να τηρήσουμε συγκεκριμένα κριτήρια για τους επενδυτές. Η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων βεβαίως και ε, συμμετέχει σε συλλογικά προγράμματα επενδύσεων όπως και άλλες τράπεζες. Και το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων που συμμετέχει σε όλες αυτές τις προσπάθειες να συμπεριλάβουμε ε, το σχέδιο Juncker για την προσθετικότητα. Το θέμα όμως της αξιολόγησης του κινδύνου είναι κάτι που ακόμα μας ε, προβληματίζει. Εάν δεν αναλάβουμε ένα συγκεκριμένο επίπεδο κινδύνου, βεβαίως δεν μπορούμε να μπούμε σε κάποια συγκεκριμένα επιχειρησιακά προγράμματα και σχέδια. Από την άλλη, κάποιοι από τους ε, τραπεζίτες οι οποίοι συμμετέχουν στα προγράμματά μας αξιολογούν τον κίνδυνο σαν όχι αρκετά υψηλό ή περισσότερο υψηλό. Βεβαίως, κάθε φορά που περνάμε μεταξύ του που περνάμε σε ένα πρόγραμμα στο οποίο συμμετέχει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, έχουμε τους σύμβουλους μας οι οποίοι μας συμβουλεύουν για το επίπεδο του κινδύνου. Πρόεδρος, έχω 12 συναδέλφους που έχουν ζητήσει το λόγο. Γι' αυτό και θα σας δώσω το λόγο στον καθένα για δύο λεπτά. Παρακαλώ πολύ να τηρήσετε το χρόνο Μιλήστε να είστε επιθαρχημένοι. Θα ξεκινήσουμε με τους σκιώδεις ομιλητές. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς επειδή θέλω να εκφράσω καταρχήν την ευχαρίστησή μου που μπορούμε να έχουμε αυτήν την συζήτηση. και ακριβώς επειδή βρισκόμαστε λίγους μήνες πριν ε, την ε, τελική απόφαση για το νέο πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο, θα ήθελα να ασχοληθούμε με κάποια λεπτά θέματα. Σήμερα βλέπουμε ότι από τη στιγμή που θα προχωρήσει το Brexit θα μας λείπουν κάποια συγκεκριμένα ποσά, κάποια δισεκατομμύρια τελικά τον χρόνο. Παραδείγματο χάρη, να σπάρουμε τον τομέα των μεταφορών. Ένα τρισεκατομμύριο για τα επόμενα 6-7 χρόνια θα μας ε, λείψει για να ολοκληρωθούν τα διευρωπαϊκά δίκτυα. Αναρωτιέμαι λοιπόν τι ακριβώς προτίθεται να κάνει η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων, ιδιαίτερα για τις πιο απομακρυσμένες περιοχές, εξόχως απομακρυσμένες περιοχές. Και δεν θα αναφερθώ σε άλλα δημοσιονομικά εργαλεία, δεν θα αναφερθώ στις εγγυήσει ή σε άλλα προϊόντα. Εσείς πώς θέλετε να προωθήσετε τα σχέδιά σας. Και αναφέρομαι εδώ και στις πιο μικρές ε, επιχειρήσεις και στις πιο απομακρυσμένες περιοχές. Επίσης, όσον αφορά το πολιετές ε, δημοσιονομικό πλαίσιο, η τράπεζά σας, πέρα από τη δική σας εμπειρογνωμοσύνη, καλείστε εδώ να υλοποιήσετε κάποιους στόχους ε, οι οποίοι ξεπερνούν το 2020. Μετά λοιπόν το Brexit, πώς βλέπετε την κάλυψη των αναγκών. Ευχαριστώ πολύ. Άλλη. Σας ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Και Αντιπρόεδρε κύριε Στούπ, αγαπητοί συνάδελφοι. Θα ήθελα καταρχάς να σας ευχαριστήσω κύριε Στούπ για την παρουσίαση των δραστηριοτήτων της ΕΤΕΠ του 2016. Ωστόσο, έχοντα υπόψη το ρόλο τη ΕΤΕΠ, δηλαδή συμβολή στην ολοκλήρωση και την κοινωνική συνοχή ε, την κοινωνική ανάπτυξη στην Ευρώπη. Έχω πολύ συγκεκριμένε ερωτήσει. Έχετε κάνει κάποιε απελευθέρωσει, αλλά εμένα μου μένουν κάποια ερωτήματα. Πρώτον, τέσσερις τομείς ε, καινοτομία, μικρομεσαίες, περιβάλλον, υποδομέ είναι οι τομείς στους οποίους ανέλαβε δραστηριότητε ε, η ΕΤΕΠ. Ποια ήταν λοιπόν, ποιο ήταν ο αντίκτυπο ήταν η κατανομή των δραστηριοτήτων ισότιμη, βέλτιστη και τι είδους σενάρια αντικτύπου και χρηματοδότηση σε διάφορες περιφέρειες σε σχέση με ΑΕΠ, και απασχόληση έχετε να μας παρουσιάσετε. Δεύτερον, χρηματοδότηση εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, 8,4 δις ευρώ σε πέντε κύριες γεωγραφικές περιοχές. Ευρωπαϊκές Συμφωνίες Ελεύθερου Εμπορίου και χώρες διεύρυνσης, χώρες προς Ανατολάς, χώρες προς Νότον και ρωτώ αν αυτό έχει γίνει σύμφωνα με τους τραπεζικούς κανόνες και αν τυχόν έχουν πληγεί ως εκ τούτου συμφέροντα των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Υπάρχει ψηλότερος κίνδυνος ως προς τις επενδύσεις εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης με τις ε, αναλύσεις σας. Για τους φορολογικούς παραδείσους ε, έχετε κάνει κάποια ανάλυση και υπάρχει κάποια συγκεκριμένη καθοδήγηση των ε, διαφόρων γραφείων σας ώστε να ακολουθούν τα επτά βήματα ε, από την υποβολή της πρότασης μέχρι την αποζημίωση ή την καταβολή των ποσών και τους κανόνες για την αποφυγή των φορολογικών παραδείσων και πού είναι οι οδηγίες. Ευχαριστώ κύριο Φλάναγκαν δύο λεπτά. Ευχαριστώ πολύ. Πολλά από αυτά που ήθελα να ρωτήσω εγώ τα έχει καλύψει ο κύριος Βάλλη. Για τις θέσεις εργασίας όμως. Εμείς ε, έχουμε κατακλειστεί από θέσεις εργασίες στην Ιρλανδία και αν αυξηθούν κι άλλο θα έχουμε ο καθένας από 4-5 δουλειές. Ε, αυτό βέβαια γιατί καμία από αυτές τις εργασίες δεν είναι αρκετή για να μπορέσει κανείς ε, να εξασφαλίσει τα προστοζή, να πληρώσει τον νίκη του, ε, να καλύψει τις καθημερινές ανάγκες του. Δουλεύουν λοιπόν σαν τα σκυλιά οι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι είναι πολύ ωφέλιμο αυτό για τον τρόπο ζωής τους. Όταν λέτε λοιπόν για 2,25 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας μέχρι το 2020, τι είδους ακριβώς τις εργασίες την υπόψη σας. Θα είναι επαρκής η κάθε μία από αυτές για να ε, επιβιώνει κανείς με αξιοπρέπεια. Και για τις επενδύσεις σχετικές με τη δασοκομεία και ιδιαίτερα με ενδιαφέρεται το θέμα των επενδύσεων αυτών στην Ιρλανδία, γιατί πολύ χρήμα είδαμε να δαπανάτε εκεί. Φαντάζομαι ότι οι επενδύσεις σας λαμβάνουν υπόψη τις ανάγκες των πολιτών, τις προδιαγραφές της ευρωπαϊκής πολιτικής για την ε, αηφορία, για τη βιοπικιλότητα. Ωστόσο, δυστυχώ, οι επενδύσει για την νοσοκομεία και διερωτώ με τι είναι ο δικό σα ρόλο εκεί, δεν βοήθησαν ούτε του πολίτε ούτε τη βιοπικιλότητα και μάλιστα έγινε δασ, ε, δασοφύτευση, ε, δέντροφύτευση σε περιοχές απόλυτα ε, ερυπωμένες, δεν έχει μείνει κάτοικος κανένας, δεν υπάρχει καμία, κανένας οικισμός ή δραστηριότητα και διαρωτώ με πώς έγιναν αυτές οι επιλογές. Το 50% της διαθέσιμης γεωργικής γης ε, τώρα έχει δεν φυτευθεί με επενδύσεις που έχετε εσείς χρηματοδοτήσει. Περιμένουμε μια ανάλυση μια έρευνα στην οποία έχουμε κινητοποιήσει. Δυτικά του άλλων δεν έχει μείνει κανένας και έχετε διώξει τους ανθρώπους ακόμη και από τις περιοχέ όπου κατοικούσαν και χρόνια πολλά. Καλή χρονιά, κυρία Πρόεδρε. Thank you, Chair. Ευχαριστώ. Και ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε που ήρθατε εδώ. Πραγματικά χαιρόμαστε ιδιαίτερα που σας ξαναβλέπουμε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Ξέρω ότι για σας το 3 είναι μαγικός αριθμός. Εγώ όμως θα ρωτήσω τέσσερα πράγματα. Πρώτον, πολύ σύντομα, ποια είναι η γνώμη σας για το γενικά υψηλό κόστος των ταμείων που διαχειρίζεται και των κονδυλίων η ΕΤΕΠ, ιδιαίτερα όταν έχουμε κοινή διαχείριση των χρηματοδοτικών μέσων. Δεύτερον, πώς ο όμιλος της ΕΤΕΠ ε, θα συνεργαστεί ε, με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ώστε να εξορθολογήσει τον αριθμό και το είδος των χρηματοδοτικών μέσων στο επόμενο ΠΔΠ. Τρίτον, τι γνώμη έχετε για τη θέση και το καθεστώς που θα ισχύσει για το Ηνωμένο Βασίλειο μετά το Brexit. Ε, είναι σαφής η κατάσταση ή είναι κάπως συγκεχημένα τα πράγματα για το τι θα συμβεί. Και Τέταρτον και τελευταίον, η, η περίοδος προβληματισμού κατά την οποία πρώην μέλη ε, του Διοικητικού Συμβολίου δεν μπορούν να κάνουν ε, λόμπι σε ε, προσωπικό και διοικητές της ΕΤΕΠ και αυτή η περίοδος ε, να παραταθεί από έξι τουλάχιστον 12 μήνες ώστε να μην έχουν πρόσβαση μετά την αποχώρηση από την ΕΤΕΠ. Αλεξάνδερ, πραγματικά χαίρομαι ιδιαίτερα που σε ξαναβλέπω. Ε, έχω τρεις ερωτήσεις ε, για κοινά θέματα φυσικά. Το πρώτο αφορά το Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων. Ε, ο προβληματισμός μας στην αρχή και το άγχος μας ήταν ότι δεν υπάρχει διάκριση μεταξύ του ΕΦΣΥ και τον, ε, το Ταμείο Συνοχής, κάποιον κονδυλίο του Ταμείου Συνοχής. Ε, Αυτά για το πρώτο εύση. Τώρα θα περάσουμε στη δεύτερη φάση. Τι διδάγματα θα αντιλήσουμε από την πρώτη φάση του εύση για να τα βελτιώσουμε στη δεύτερη του φάση. Δεύτερη ερώτηση. Αφορά και πάλι την κατάσταση του Ηνωμένου Βασιλείου, το καθεστώ του μετά τον Brexit. Ε, σίγουρα ε, σεβαστή η απόφαση, παρόλο που ε, Μα θλίβει και λυπόμαστε γι' αυτό και δεν ξέρουμε πώς θα διαμορφωθεί η μελλοντική σχέση με την ε, Ευρωπαϊκή Ένωση. Ποια είναι η νομική βάση για τη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στην ε, τράπεζα ΕΤΕΠ και στο μέλλον ε, υπάρχει δυνατότητα να συνεχίσει να, παραμένει, το Ηνωμένο Βασίλειο μέλος της ΕΤΕΠ. Βλέπετε κάποια, κάποιο τρόπο για να διασφαλιστεί. Ο κύριος Λιμπεράτσκι για δύο λεπτά. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αγαπητέ Αντιπρόεδρε Αλεξάνδρε Στούπ, καλώς ήρθατε και πάλι στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Συμφωνώ μαζί σας ότι ε, οι επιδόσεις και ο ρόλος σας ε, είναι θετικός. Συμφωνώ μαζί σας και δεν θα σταθώ σε αυτό. Εμένα με ενδιαφέρει το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατηγικών Επενδύσεων, το ΕΦΣΥ, η ΕΤΣΕ, σε ό,τι αφορά τη γεωγραφική κατανομή και την ε, προσπάθεια να βοηθήσει τις λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες. Είχαμε πρόσφατα μία σχετική δημόσια ακρόαση και θέλουμε να εντρυφήσουμε στο θέμα αυτό για να αντιληφθούμε τους μηχανισμούς του ΕΦΣΥ πώς μπορεί να στηρίξει τις ε, λιγότερο ανεπτυγμένες περιφέρειες για να καλύψουν το χαμένο έδαφος. Και μάλιστα ε, στο τέλος της δημόσιας ακρόασης ε, ακούσαμε κάποιες συστάσεις. Πώς μπορούμε λοιπόν να βελτιώσουμε την συνδρομή του ΕΦΣΥ ε, εν ώψη και του επόμενου πολίτους δημοσιονομικού πλαισίου γιατί θα δημιουργήσει ένα διαφορετικό περιβάλλον και λόγω του Brexit. Και κατά πάσα πιθανότητα το νέο επιδελταπή ίσως αυξήσει τις επενδύσεις ε, και εστιαστεί σε μια επαναβιομηχανοποίηση. Και να το δούμε στη συνάφεια και με το Ταμείο Συνοχής ε, και άλλα ταμεία που ίσως ε, συνδυαστούν με το ΕΦΣΥ για να ανέλθουμε στα 500 δις εκατομμύρια επενδύσεων. Ευχαριστώ. Κύριο Σαλαφράγκα. Ευχαριστώ, ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε και εγώ θα ήθελα να καλωσορίσω τον ε, παλιό μας συνάδελφο Αλεξάνδερ Στούπ και να τον ευχαριστήσω για τις πληροφορίες που μας έδωσε ε, για την έκθεση της τράπεζας για τις εργασίες του 2016. Πολύ εντυπωσιακή σημαντικό το έργο, είναι η πιο σημαντική τράπεζα του κόσμου ίσως και μάλιστα είχε πάνω από 400 ε, δισεκατομμύρια στο, στην αγορά κεφαλαίων και μας είπε για 25 ε, εκατομμύρια ε, ανθρώπους που έχουν καλύτερη πρόσβαση σε υδροδότηση, 20 εκατομμύρια σε καλύτερη, καλύτερο εξοπλισμό, 10 εκατομμύρια έχουν πια πρόσβαση σε καλύτερες υγειονομικέ εγκαταστάσεις χάρη στα έργα και τα προγράμματα της ΕΤΕΠ. Έχω τρει ερωτήσεις όμως. Όπω ο κύριος Βάλλη και άλλοι, θεωρώ ότι το Ευρωπαϊκό Ταμείο Στρατικών Επενδύσεων μέχρι στιγμής έχει κινητοποιήσει μόνο 163 δισεκατομμύρια, τα μισά δηλαδή από ό,τι είχε προβλέψει να προσελκύσει, που ήταν περίπου 300 δισεκατομμύρια. Είμαστε περίπου στο 50% των στόχων. Φυσικά δεν έχει εκπνεύσει ακόμη η περίοδος των προβλέψεων, αλλά θα ήθελα να μου πείτε ε, πώς ε, πρόκειται να υλοποιήσουμε αυτό το στόχο και σε τι ρυθμό ε, βαδίζουμε. Σε ό,τι αφορά τις τρίτες χώρες, 980 εκατομμύρια αφιερώσετε στις χώρες Τη Ασία και τη Λατινική Αμερική. Ε, Ποιο ήταν ο επιμερισμός μεταξύ των δύο περιοχών τη Ασία και τη Λατίνική Αμερική, και ποιε είναι οι προβλέψει για το επόμενο έτος. Και τελευταία ερώτηση, κυρία Πρόεδρε. Ποια είναι η θέση της ΕΤΕΠ σε ό,τι αφορά τα φιλοπεριβαλλοντικά ομόλογα ή τα ομόλογα με κλιματική συνείδηση. Γιατί 380 ε, δισεκατομμύρια ήταν οι επενδύσεις φέτος και η ιδιαιτερότητα είναι τα 21 χρόνια διάρκεια. Ποια είναι η θέση της ΕΤΕΠ σε σχέση με τέτοια πράσινα ομόλογα. Ο κ. Σέλερ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Στούπ. Χαίρομαι που σε βλέπω πάλι εδώ μεταξύ μου. Και καταρχήν θα ήθελα να πω πόσο εκτιμώ την εργασία της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων. Όσον αφορά όμως την εύση του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, Βεβαίως ε, υπάρχει η συμμετοχή σε όλη αυτή την ε, επενδυτική δραστηριότητα, σε προγράμματα και βλέπουμε ότι συνεργάζεστε όλο και περισσότερο με τις τράπεζες προώθησης της EPB. Ε, Ήθελα να μου πείτε πώς η αξιολόγηση του κινδύνου η συμμετοχή σας σε αυτά τα προγράμματα μπορεί να συμβαδίζει και πώς ελέγχεται ότι οι επενδύσεις και η χρηματοδότηση των υπόλοιπων ποσών ε, γίνονται από άλλους φορείς. Πώς δηλαδή η χρήση των κονδυλίων και των ποσών που επενδύονται ελέγχονται, αν ε, δίνονται ποσά αρκετά για θέματα ενεργειακής μετάβασης. Σε εμά αυτό είναι ένα πάρα πολύ σημαντικό θέμα και βεβαίως ε, μπορεί αυτό να γίνει και από κάποια ποσά τα οποία μέχρι τώρα δινόταν σε επιδοτήσεις και τα οποία δεν έχουν ε, απορροφηθεί παραδείγματος χάρη. Θα ήθελα επίσης να μου πείτε γιατί εμείς θέλουμε σαν Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να συνεχίσουμε να παίζουμε το ρόλο που παίζουμε στον έλεγχο αυτών των ε, επενδύσεων. Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι τα ποσά αυτά θα συνεχίσουν να επενδύονται σωστά και επίσης όσον αφορά τις αποζημιώσεις θα ήθελα να μου πείτε και τις επιστροφές ποσών θα ήθελα να μου πείτε τι ακριβώς προγραμματίζετε να κάνετε. Και το θέμα της Αφρικής επίσης με ενδιαφέρει. Ευχαριστώ πολύ. Έχω μια πολύ σύντομη ερώτηση, κύριε Αντιπρόεδρε, θα ήθελα να μιλήσουμε για το θέμα των κινδύνων. Ποιοι είναι οι δικοί σας τρόποι αξιολόγησης του κινδύνου, τα κριτήριά σας και όσον αφορά την σωστή χρήση των ποσών, των κονδυλίων. Μπορείτε να μας πείτε κάτι. Βεβαίως δεν θέλω να αναφερθείτε σε συγκεκριμένα προγράμματα, αλλά για το 2016 μας δώσατε κάποια στοιχεία για τα συνολικά ποσά που δώσετε σε δάνεια. Θα ήθελα να μου πείτε τι γίνεται με τα επόμενα χρόνια. Ευχαριστώ πολύ. Η κυρία Γιάλα Σέντερ, ευχαριστώ και καλώς ήρθατε και από μένα κύριε Στούπ. Εκπροσωπώ εδώ τον κύριο Πυρίνσκι που χρειάστηκε να μεταβεί στην Επιτροπή Απασχόλησης. Εκ μέρους του θα ήθελα να υποβάλω κάποιες ερωτήσεις. Η έκθεση της ΕΤΕΠ γνωρίζετε ότι δεν είναι αρκετά περιεκτική γιατί η εκθέση δραστηριοτήτων ε, των ε, επιχειρήσεων της ΕΤΕΠ και εντός και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης δίνουν πιο διεξοδικές ε, πληροφορίες σε σχέση με την ετήσια έκθεση δραστηριοτήτων που περισσότερο έχει διαφημιστικό επικοινωνιακό χαρακτήρα παρά αναλυτικό. Επανειλημμένως ε, ζητήσαμε μια σφαιρική περιεκτική και πιο διεξοδική έκθεση. Πότε επιτέλους θα λάβουμε μια τέτοια ολοκληρωμένη περιεκτική έκθεση που μας είναι απαραίτητη και για το δικό μας κοινοβουλευτικό έργο. Δεύτερον, σε ό,τι αφορά τον ε, γεωγραφικό επιμερισμό, τη γεωγραφική κατανομή. Το 2016 διαπιστώνουμε ότι τρεις χώρες, η Βουλγαρία, η Κροατία και η Λετωνία, δεν έχουν ε, λάβει ούτε ένα δάνειο αυτό είναι εντυπωσιακό. Ενώ άλλες χώρες όπως η Λετωνία, η Μάλτα και μία τρίτη δεν είχε πρόσβαση ούτε σε εγγυήσεις ούτε σε άλλο είδους ε, χρηματοδοτικών μέσων. Γιατί λοιπόν οι χώρες αυτές δεν κατάφεραν να υποφεληθούν από την συμβουλή της ΕΤΕΠ και να λάβουν κάποια κονδύλια για προγράμματα. Επίσης, ε, τι γίνεται με τις επενδύσεις υπέρ της συνοχής στην Ευρωπαϊκή Ένωση σε σχέση με το 2015. Στην περίπτωση του ΕΦΣΙ, του Ευρωπαϊκού Ταμείου Στρατηγικών Επενδύσεων, φαίνεται ότι όχι μόνο υπάρχει πρόβλημα στην γεωγραφική κατανομή, αλλά και στην ε, τομεακή κατανομή, την κλαδική κατανομή. Γιατί σε κάποιου τομείς όπως ε, στις κοινωνικέ επενδύσεις, εκεί το ΕΕ δεν εμφανίζεται να προσφέρει στοιχεία. Επίσης, αναθεώρηση του θετολογικού κώδικα, του κώδικα συμπεριφορά, κλπ. Ναι, ναι, συγγνώμη, αλλά θα τελειώσετε τώρα, κύριος Δεγιόγκο. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο Στούπ για την παρουσίασή του και για την ε, έμφαση στην διαφάνεια. Η αναθεώρηση του μηχανισμού προσφυγών της τράπεζας με ενδιαφέρει ιδιαίτερος στο πλαίσιο των ε, διαβουλεύσεων ε, με το κοινό βλέπουμε ότι υπάρχουν ιδιαίτερες επισημάνεις σε σχέση με την προσβασιμότητα σε αναφορές και διαμαρτυρίες ένσταση των πολιτών. Κανονικά θα πρέπει να δώσετε μια απάντηση σε αυτό, αλλά δεν βλέπω τίποτα και φαντάζομαι ότι είναι ένα σημαντικό κομμάτι της διαφάνειας να δοθούν και απαντήσεις. Επίσης, Ένα δώρο 400 εκατομμυρίων ευρώ προς τη Volkswagen. Ανέλαβε η Όλαφ δραστηριότητα νομίζω και επελήφθη να μελετήσει το θέμα αυτό, όπως άλλωστε και το θέμα των εκπομπών καυσαζερίων. Θα θέλαμε λοιπόν να μας πείτε Πού βρίσκεται αυτό στην έκθεσή σας ή μήπω η ΕΤΕΠ μόνο με την, στην όλα φλογοδοτή και μετά γίνεται αυτή η, ε, η μετάδοση των πληροφοριών. Μπορείτε να μας διαβεβαιώσετε ότι θα υπάρξουν περαιτέρω ε, προβλήματα στο μέλλον. Η Πρόεδρος θέλω και εγώ να πω δύο λόγια. Είναι σχετικά ασφαλές το σύστημα, 316 εκατομμύρια από τη διαχείριση των διαρθρωτικών ταμείων και από δημοσιονομικά μέσα. Επομένως δεν υπάρχει θέμα να αναζητηθεί από που είναι ξεκάθαρο για όλους. Για τον κύριο Βάλη. Ε, δίνουμε ε, σαφή απάντηση στο γεγονός ότι είναι η ΕΤΕΠ ε, εκείνη η οποία παρακολουθεί τον τρόπο με τον οποίο οι ιδιωτικές τράπεζες προβαίνουν σε επενδύσεις και βέβαια και των ιδιωτικών επενδύσεων γιατί πιστεύω ότι αυτές οι ιδιωτικές επενδύσεις οδηγούν και σε προσέλκυση ιδιωτικών κονδυλίων από ιδιωτικές ε, εθνικές πηγές, πόσο, τι ποσό λοιπόν ιδιωτικών κονδυλίων και πόσους νέους συνεργάτες προσλάβατε το 2016 και μετά το 2017 για τη διαχείριση όλων αυτών και τώρα έχετε εσείς το λόγο. Ευχαριστώ Πρόεδρε. για το ευρύ φάσμα των ερωτήσεων και θα κάνω ό,τι μπορώ για να δώσω απαντήσεις στις περισσότερες από αυτές τουλάχιστον. Για να είμαστε πιο σαφείς θα αναφερθώ στο κάθε χωριστά, στην κάθε ερώτηση χωριστά και αν τυχόν κάτι παράλληψα παρακαλώ να μου το επισημάνετε. Ο κύριος Νόβακομ για την προαγωγή των προϊόντων μας και την επίτευξη των στόχων το 2020. Δεν νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα. Μάλλον νομίζω ότι είχαμε πρόβλημα επικοινωνιακό, δηλαδή δεν προβάλαμε αρκετά αυτό που κάναμε στο κοινό. Η επικοινωνιακή πολιτική της τράπεζας που έχει πίσω τις έξι χρόνια όταν ε, ε, είναι ότι όταν ε, δεν μας ε, ακούνε στα μέσα μαζικής ενημέρωση. Αν δεν εμφανίζεται το όνομά μας στα μέσα Μαζική ενημέρωση, είναι καλό. Αυτή ήταν γενικά η τακτική όλα αυτά τα χρόνια. Δεν κάνουμε τίποτε για να διαφημιζόμαστε, δεν προβαλόμαστε. Θέλουμε οι δράσεις μας να μιλούν για μας και νομίζω ότι με το έτσι μπορέσαμε να πάρουμε μια σαφή όθηση προς την κατεύθυνση αυτή. Επίσης, στην ΕΤΕΠ κάποιοι αντιπρόεδροι έχουμε ε, και πολιτικό υπόβαθρο ε, παρελθόν ε, ενασχόληση με την πολιτική και εμείς ίσως θα θέλαμε να ενισχύσουμε το πολιτικό μήνυμα αλλά βέβαια υπάρχουν και οι εντό τεχνοκράτες αντιπρόεδροι που δεν το επιθυμούν αυτόν. Αυτό. Για το 2020 νομίζω ότι μεγάλο κομμάτι της δουλειάς θα είναι το, 2000, είναι το πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που και σας απασχολεί ασφαλώς για το πολιετές δημοσιονομικό πλαίσιο λοιπόν και βεβαίως η τράπεζά μας θα διατυπώσει τις θέσεις της, θα τις υποβάλει το Φεβρουάριο. Θα υπάρξει μείωση στις ενισχύσεις και φαντάζομαι ότι η πρόταση της Επιτροπής θα μπορούσε να προσφέρει σε 10% μόνο δημοσιονομικά μέσα και δημοσιονομικές εγγυήσεις ε, ποσά σε σχέση με τον τωρινό προπολογισμό μόνο το 10% και μετά θα πρέπει οι τράπεζε να καλύψουν το υπόλοιπο. Και αυτό πια θα είναι η δική μα δουλειά. Γιατί, θα σα δώσω ένα παράδειγμα, το 10% εάν είναι 15 δισεκατομμύρια, η μόχλευσή του είναι τριπλάσια, δηλαδή 45 δισεκατομμύρια λειτουργικού όγκου, επιχειρησιακού όγκου για μας και εδώ βεβαίως θα έρθω και στη δική σας την ερώτηση για την επάντρωση γιατί θα πρέπει βεβαίως και εμείς να είμαστε θέση να το διαχειριστούμε. Για τον κύριο Αλή που είχε μια-δυο ερωτήσεις. Συνέπειση επί του ΑΕΠ και της απασχόλησης και εξωτερικών επενδύσεων, επενδύσεων εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το είπα ήδη στην ε, εισαγωγική μου παρέμβαση η απόδοση της δράσεως της ΕΤΕΠ οδήγησε σε 2,25 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας, 2,3 επί του ΑΕΠ έως το 2020, τα 2,25 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας είναι για το 2015 και το 2016. Για το δεύτερο θέμα τώρα, για το πώς προσαρμοζόμαστε στους κανόνες, η δεύτερη ερώτηση του κυρίου Αρλή είναι πραγματικά απόλυτα αυστηρή η εκτέλεση του καθήκοντος επιμέλειας της τράπεζας και εγώ ε, μπορεί να έχω ένα, ένα υπόβαθρο και ένα ιστορικό ενασχόληση με την πολιτική και τα οικονομικά. Έχω να σας πω όμως το εξής ότι υπάρχει ένα τμήμα Ε, υπεύθυνων για τη χορήγηση δανείων ή επιχειρησιακών, επιχειρησιακό τμήμα που εξετάζει όλες τις προϋποθέσεις. Μετά πάμε στη διαχείριση του έργου που επίσης εξετάζει τις προϋποθέσεις και την τήρησή τους. Μετά έχουμε τους δικηγόρους, μετά έχουμε τους ε, τα στελέχη τα ειδικά για την ανάλυση κινδύνου και μετά έχουμε τα στελέχη ε, που ασχολούνται με την χορήγηση του δανείου. Αυτό λοιπόν γίνεται κάθε φορά πριν από την ε, χορήγηση δανείου από ένα δημοσιονομικό μέσο. Και είναι πάρα πολύ αυστηρό ο έλεγχο. Κάθε φορά που κάποιο καταφέρει να τον περάσει και να εγκριθεί το έργο του, αξίζει συγχαρητηρίων. Ε, η διαφορά σε σχέση με τι κοινέ τράπεζε σε εμά είναι ότι όταν έρχεται ένα έργο, ένα αίτημα για δάνειο, ένα δημοσιονομικό μέσο, δεν το εξετάζουν μόνο οι οικονομολόγοι. Υπάρχουν οικονομολόγοι, υπάρχουν οι μηχανικοί, υπάρχουν οι επιστήμονες οι γιατροί, οι δικηγόροι που θα το εξετάσουν ως προς την βιωσιμότητά του και φυσικά αυτό ε, εξηγεί και γιατί έχουμε το χαμηλότερο ποστό μη εξυπηρετούμενων ε, δανείων. Ο κύριος ε, Φλάναγκαν έκανε μια πολύ ενδιαφέρουσα παρατήρηση για τη δημιουργία θέσεων εργασία. Δεν μπορώ να σας δώσω απάντηση για το ποιε θα είναι οι 2,25 δισεκατομμύρια θέσεις εργασίας. Μπορούμε να συζητήσουμε και τη ρομποτοποίηση, την αυτοματοποίηση, ε, την τεχνητή νοημοσύνη, τη τρισδιάστατη εκτύπωση, την ψηφιοποίηση και τις συνέπειές τους στις θέσεις εργασίας στο μέλλον. Αλλά αυτό δεν μπορούμε εμείς να το ορίσουμε. Ε, εμείς είμαστε τράπεζα και εμείς ε, καλούμε τον κόσμο να κοιτάξει το καλό που μπορούμε να προσφέρουμε ως τράπεζα και επίσης πιστεύω ότι λόγω των πολύ αυστηρών συνθήκων που αντιμετωπίζουμε και των όρων ε, για τη δουλειά μας προσφέρουμε πολλά χωρίς να μπορώ να αποκλείσω κάθε πρόβλημα για την δασοκομεία παραδείγματι έχουμε 300 που διαχειρίζονται τέτοιου είδους εγχειρήματα στο προσωπικό μας κάνουμε ό,τι μπορούμε εν πάση περιπτώσει Ο κύριο Σάουαρμα επίσης έκανε πολύ ενδιαφέρουσε ε, ερωτήσεις ε, το υψηλό κόστος και τα τέλη ε, στην υλοποίηση των δημοσιονομικών μέσων της ΕΤΕΠ. Σε αυτό θα απαντήσω πρώτα ότι πολλές από τις κοινέ τράπεζες δεν μας συμπαθούν γιατί έχουμε χαμηλά τέλη, έχουμε τριπλό αλφα, λίγες τράπεζες μας φτάνουν από τα 28 κράτη-μέλη. Οπότε έχω να απαντήσω το εξή. Ότι ναι, μπορεί να λέτε ότι είναι ακριβά τα τέλη αλλά στην πραγματικότητα είμαστε φθηνότεροι από πολλά χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Επίση, έχουμε διαχείριση σε περιφερειακό επίπεδο, σε κοινό επίπεδο των κονδυλίων και όποτε υπάρχει αύξηση ε, τιμών σε ένα ταμείο, ε, σε ένα κονδύλιο που μπορεί εμείς να συμμετέχουμε, αυτό αυτόματα αυξάνει και τα τέλη. Και ταυτόχρονα αντιμετωπίζουμε και το θέμα ενός ανώτατου επίπεδου που προσδιορίζει τιμές και μετά από αυτό δεν μπορούν να αυξηθούν. Σας διαβεβαίω πάντως ότι είμαστε φθηνοί για αυτό που προσφέρουμε. Επίση, υπήρξε μια ερώτηση για το αν θα συνεργαστούμε ενεργά με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ω προ τον εξορθολογισμό των ε, μέσων. Η απάντησή μου είναι θετική, ναι ώψη και του 2020 οπωσδήποτε. Ταυτόχρονα όμω θέλω να, επισημάνω ότι ακριβώ επειδή η Επιτροπή μα έχει ζητήσει να μειώσουμε κάποια μέσα του έτσι, ε, έχουμε μια συσσόρευση, τα εξετάζω, δεν είμαι οικονομολόγος, ε, κοιτώ τα δημοσιονομικά με μέσα της, τις οικονομικές υπηρεσίες του ΣΥΠΗΝ και τις δυνατότητες που προσφέρονται και βέβαια υπάρχουν πάρα πολλά μέσα. Προσπαθούμε να τα εξορθολογήσουμε όλα, να τα κάνουμε πιο, πιο απλά, αλλά ταυτόχρονα είμαστε υποχρεωμένοι και να βρούμε τη λύση μέσα από την απλοποίηση. Και βεβαίως στο ερώτημα το σχετικό με το Brexit για τον κύριο Σάουαρμα και τον κύριο Ashworth Πιστεύω ότι η συμφωνία της 7ης Δεκεμβρίου έλυσε το θέμα των σχέσεων μεταξύ Ευρωπαϊκού, ε, Ευρωπαϊκής Τράπεζας ε, Επενδύσεων και Ηνωμένου Βασιλείου με 60% συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου εκ των οποίων το ίμιση πηγαίνει σε αυτό που καλύπτεται ε, προκαταβολικά και το υπόλοιπο ποσό που θα είναι το ποσό εγγυήσεως όπως τα λέγαμε το πρώτο είναι το 3,5 δις το καταβεβλημένο ποσό, θα πρέπει να το επαληθεύσουμε βεβαίω. Και αυτό στα δεκαετία θα επιστραφεί. Από την ημέρα δηλαδή τη συμφωνία, όταν περάσουν 12 χρόνια, θα επιστραφεί σε δόσει των 300 εκατομμυρίων ευρώ ποσό μετρητή δηλαδή που κατατίθεται και επιστρέφεται 12 χρόνια γιατί τόση είναι και η κύκλη των ε, δανείων, κάποιων δανείων. Το ποσό εγγύησεως 35 με 36 δισεκατομμύρια θα μπει σε ένα ε, ταμείο εγγύησεως και θα παρακολουθεί την εξέλιξη και την ορίμανση των δανείων. Γιατί έχουμε δάνεια και 30-40 ετών στο Ηνωμένο Βασίλειο. Νομικό τώρα ζήτημα. Το Ηνωμένο Βασίλειο παραμένει να μέλος, μπορεί να παραμείνει μέλος της ΕΤΕΠ. Όχι. Αυτό προβλέπει η συνθήκη, αυτό προβλέπουν οι κανονισμοί. Την, ε, της ΕΤΕΠ κύριοι και οι ιδιοκτήτες είναι τα κράτη-μέλη. Διαφορετικό το θέμα του Ευρωπαϊκού Νομισματικού Ταμείου, αλλά για την ΕΤΕΠ το Ηνωμένο Βασίλειο δεν μπορεί να παραμείνει μέλος. Βεβαίω θέλουμε να συνεχίσουμε τη συνεργασία, καμιά αντίρρηση σε αυτό. Είναι μεγάλο το θέμα, όπω μεγάλο θέμα βέβαια προκύπτει και για την δραστηριότητα τη τράπεζα. Για μα πρόκειται και απόλυτα ασφαλώ. Δεν θα θέλαμε να χάσουμε έναν από του κυρίου μετόχου μα, αλλά έτσι είναι τα πράγματα και πρέπει να τα αντιμετωπίσουμε. Και μετά, περίοδος αναλογισμού που αναφέρατε, ε, δεν μπορώ να σας απαντήσω. Δεν γνωρίζω το θέμα τόσο καλά. Εάν εννοείται για το προσωπικό, για τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου, των ε, διευθυντών δηλαδή που προέρχονται από τα κράτη-μέλη, από 6-12 μήνες, δεν ξέρω, μπορεί κανείς να το εξετάσει, αλλά δεν ε, ξέρω πώς λειτουργεί το σύστημα. Για τους αντιπροέδρους ναι έχω απάντηση, αλλά όχι για τους υπαλλήλου. Προσθετικότητα του κυρίου Ashworth. Φαντάζομαι να απάντησα τα διδάγματα από το πρώτο έτσι και από το δεύτερο έτσι, τα τέσσερα σημεία πάνω στα οποία θέλουμε να δώσουμε περισσότερη έμφαση, οι συμβιβασμοί μεταξύ Κοινοβουλίου, Επιτροπής, κράτων μελών ε, για το έτσι ασφαλώς θα γίνουν σεβαστά. Και για τον κύριο Λιμπεράτσκι τώρα, γεωγραφική ανάλυση. Ξέρετε, έχω τα στοιχεία του 2017 για την κατανομή θα δημοσιευθούν άλλωστε σήμερα, από ό,τι γνωρίζω, στο ιστοσελίδα μας. Δεν πιστεύω να διαφέρουν πολύ από τα στοιχεία του 2016. Σας δώσω όμως κάποιες, σε κάποιες αντρές γραμμές. Η Πολωνία, παραδείγματι, παρουσιάζει εδώ ιδιαίτερο ενδιαφέρον, η ΕΤΕΠ έχει χρηματοδότηση στην Πολωνία 5,4 δις το 2017. Για άλλες μεγάλες χώρες μπορώ να σας αναφέρω η Ισπανία. 10,8 δις. Οι κάτω 2,6 δις. Η Φινλανδία 1,6 δις. Η Γερμανία 7,25 δις και ούτω καθεξής. Αλλά πραγματικά εμένα με ενδιαφέρει άλλο στοιχείο. Είναι η χρηματοδότηση αναχώρα ως ποσοστό επί του ΑΕΠ με πρώτη την Κύπρο, δεύτερη την Ελλάδα, τρίτη την Κροατία, μετά την Πολωνία, την Ρουμανία, την Πορτογαλία, την Ισπανία, την Εσθονία, την Ιταλία και την Ουγγαρία και άλλες μετά. Φυσικά αυτό μπορεί να κυμαίνεται από χρόνο σε χρόνο, αναλόγως ε, της χρονιάς. Δύο δίσφαιροι πίν ε, κάποια στιγμή στην ε, Ισπανία και έτσι έρχεται σε υψηλό επίπεδο η Ισπανία. Κάποιες χώρες ακούστηκε δεν ε, δέχονται καμία επένδυση. Όχι, δεν ισχύει αυτό. Όλες οι χώρες είναι κομμάτι της, ε, του ΕΤΣΕ, καλύπτονται από το ΕΤΣΕ και βέβαια τις ε, επενδύσεις της ΕΤΕΠ για το 2017. Και για το ΕΤΣΕ μια ερώτηση του κυρίου Σαλαφράγκα. τα στοιχεία δείχνουν μια καλύτερη εικόνα από ό,τι αναφέρετε εσείς. 256 δις αυτή τη στιγμή με 82% ποσοστό από τα 315 δις. Το δικό μας επιχειρηματικό σχέδιο, το λεγόμενο COP, θα μας επιτρέψει να καλύψουμε το όριο αυτό. Για το έτσι συγκεκριμένα, όταν έλεγα νωρίτερα ότι θα πρέπει να γίνει πιο ε, ε επιφυλακτικό απέναντι στον κίνδυνο. Ήταν λάθο όρο που χρησιμοποίησα. Έπρεπε να πω αντιθέτω ότι θα πρέπει να γίνει πιο ρήψο κίνδυνο. Ε, έχουμε χρησιμοποιήσει για τη διεύρυνση και 7, 1,6, Ανατολική Γειτονία 1,88, Μεσόγειος 1,96, Ακαίος Αφρική 1,47, αφρικη Νότια Νότιο-Ανατολική Ασία, Λατινική Αμερική. 1,99 δις είναι η κατανομή των ποσών ε, που ζητήσατε εσείς νωρίτερα. Νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικό να γίνει εξορθολογισμός της ε, χρηματοδότηση του τομείου αυτό για να είμαστε και πιο αποτελεσματικοί. Μιλήσατε για πράσινα ομόλογα. Συνεχίζουμε. Συνεχίζουμε με την έκστρατη ε, αυτή έκδοσης. Και στις τελευταίες ερωτήσεις... Τσέλερ, ποιος παρακολουθεί και επιτηρεί τις επενδύσεις ε, τρίτων. Έχουμε ένα τμήμα συμμόρφωσης που ονομάζεται ΟΚΟΚΟ, OCCO, αυτή είναι η διολεκτός μας, το οποίο με ευξημένη ε, επιμέλεια στη συνεργασία και με τους δικηγόρους και με τους ε, επιμελητές των έργων, των δανείων κτλ. παρακολουθεί την τήρηση. Δεν είναι ότι είναι όλα άψογα και τέλεια. Από τα δέκα έργα τα δύο πάντα θα έχουν κάποιο ζήτημα συμμόρφωσης που θα συσχετίζεται και με την επιτήρηση διότι εμείς βεβαίως ιδιαίτερα Ανησυχούμε να μην πληγεί το κύρος μας και η αξιοπιστία, η μας, ο λεγόμενος ψυχολογικός κίνητρος. Γι' αυτό δεν θέλουμε να είναι κάποιο σχέδιο ε, εκτεθειμένο σε επικρίσεις ή μομφές. Γι' αυτό είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί στην ε, ε παρακολούθηση για τον κύριο Κόρν και τα κριτήρια κινδύνου. Μπορεί τα κριτήρια μας να είναι τα ίδια με άλλες τις κοινέ τράπεζες, αλλά το πρώτο σημείο διαφοράς είναι ότι εμείς δεν είμαστε κερδοσκοπική τράπεζα, ενώ οι άλλες είναι ε, κερδοσκοπικές και άσως εκ του αναλαμβάνουν περισσότερους κινδύνους. Επίσης, η διαδικασία ε, δέουσας επιμέλειας είναι εκ των πιο, αν όχι ή πλέον αυστηρή στον κόσμο, γι' αυτό έχουμε και το χαμηλότερο ποσοστό ε, μη εξυπηρετούμενων δανείων με 0,3% κατά μέσο πέρσι μόνο, κατά μέσο όρο 0,4%, ποσοστό που δεν έχει καμία τράπεζα στον κόσμο. Τι θα γίνει στη συνέχεια δεν ξέρω, μπορεί να υπάρξουν άλλα μια εξυπηρετούμενα ή περισσότερα μια εξυπηρετούμενα δάνεια. Ε, νομίζω ότι το 717 ήταν μόνο 26 σε αυτή τη χρονική περίοδο. Ε, όπως και να έχει, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν πρόκειται να πάρουμε ποτέ τα λεφτά μας πίσω. Απλώς ε, ανεβάζουμε κόκκινο σημαία και αρχίζουμε και μελετούμε με ιδιαίτερη προσοχή και παρακολουθούμε την εξέλιξη του δανείου αυτού και την εξυπηρέτησή του. Κυρία Αγιάλα Σέντερ, με ρωτήσατε εκ μέρους του κύριου Περίσκη το θέμα της γεωγραφικής κατανομής, ε, τις ολοκληρωμένες εκθέσεις θα επανέλθω στο θέμα αυτό. Επίσης, ο κύριος Ντεχιόγκ μίλησε για την αναθεώρηση του, του κανονισμού για την υποβολή αιτιάσεων. Ε, μόλις ε, συζήτησα αυτό το θέμα με, τον αρμόδιο, με το αρμόδιο τμήμα και έχουμε περίπου 5.000 ερωτήσεις ή παράπονα που έχουν υποβληθεί στο αρμόδιο τμήμα και ε, το Φεβρουάριο του 2018 θα συζητήσουμε στην ε, Διοικητική Επιτροπή όπως αναφέρεται στις δημόσιες διαβουλεύσεις για το 2017. Και θα εγκύψω στο συγκεκριμένο θέμα μέσω μόλις ε, ε, επιστρέψω και ελπίζω να σας δώσω απάντηση. Γιατί μερικές φορές έχουμε κάποιες καθυστερήσεις για το θέμα της Volkswagen. Πολύ ευχαρίστως να σας στείλω γραπτό στην απάντησή μου. Όντως ήταν λεπτό το θέμα και ευαίσθητο και επειδή μπήκε και δημοσίως το θέμα, θα ήθελα να είμαι ακριβή στην απάντησή μου. Θα τη στείλω γραπτός. Και κυρία Πρόεδρε, λυπάμαι που μακρηγόρησα κάπως. Το θέμα των εθνικών τραπεζών πρόθεσης είναι πολύ σημαντικό ε, και το θέμα των εθνικών τραπεζών πρόθεσης ε, ήταν καταρχήν το ΕΦΣ ήταν καλό για μας γιατί συνεργαστήκαμε με τις εθνικές τράπεζες πρόθεσης δεν υπήρξε συναγωνισμός μεταξύ μας και ο πρόεδρος Βέρνερ Χόιερ από ιδιαίτερη σημασία στι εθνικέ τράπεζε πρόθεση και συνεργάζεται στενά μαζί τους. Και έχουμε 25 μνημόνια συνεννόησης με διάφορες Εθνικές τράπεζε πρόθεση, ε, που έχουν διαφορετικά χαρακτηριστικά σε κάθε χώρα. Μερικές χώρες δεν έχουν καν τέτοιες. αλλά το πιο σημαντικό είναι ε, στο ΠΔΠ. Όσοι ασχολούνται με το πολιτές δημοσιονομικό πλαίσιο, ε, αν όπως προτείνει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, καταλήξουμε σε ένα νέο ταμείο και από αυτό αρχίζουμε να χρησιμοποιούμε με μεγαλύτερο αριθμό χρηματοδοτικών μέσων και δημοσιονομικών εγγύσεων, τότε η ΕΤΕΠ είναι πάνω από το πεδίο ισότιμου ανταγωνισμού, γιατί η συνθήκη της αναθέτει το καθήκον να εφαρμόσει καινοτομίε και θα πρέπει να βρούμε διάβλους για στενότερη συνεργασία με τις Εθνικές Τράπεζες Πρόθεσης και είμαι σίγουρος ότι θα το καταφέρουμε. Τώρα για τα ιδιωτικά κονδύλια σε σχέση με τα δημόσια, δεν έχω συγκεκριμένα νούμερα. Πάντω σίγουρα προσελκύουμε επενδύσει και από τον ιδιωτικό τομέα, αλλά τα ακριβή στοιχεία θα σα τα δώσω αργότερα. Για το νέο προσωπικό, θα γνωρίζετε, καταρχήν όταν ξεκίνησε το ΕΦΣΥ, είχαμε περίπου 2.500 υπαλλήλου ε, για τα γραφεία μα ανά τον κόσμο αλλά και κυρίω στην Ευρώπη. Τώρα έχουμε φτάσει στου 4.000 υπαλλήλου. και μάλιστα αυτή τη στιγμή έχουμε παγώσει τι προσλήψει για πολλούς και διάφορους λόγους δεν μπορούμε να προσλάβουμε και άλλους. Πάντως η αλήθεια είναι ότι όσο αυξάνονται ε, οι αρμοδιότητές μας και οι επιχειρήσεις μας, τόσο περισσότερο προσωπικό θα χρειαζόμαστε. Και είναι ενδιαφέρον το θεσμικό αυτό μας όργανο, η ΕΔΕΠ, γιατί έχει πολλούς νέους υπαλλήλους. Εγώ πέρασα σχεδόν από όλα τα κοινοτικά θεσμικά όργανα και μερικές φορές ε, κάποιος όταν ξεκινάει σε ένα κοινοτικό θεσμικό όργανο παραμένει σε αυτό. Ε, εμείς στο προσωπικό μας έχουμε δηλωμένη δέσμευση να παραμείνουν ε, για πολλά χρόνια. Αλλά τώρα έχουμε ένα νέο σύστημα με τετραετή συμβάσεις και προσελκύουμε πολλούς νέους. Αλλά τα ακριβή στοιχεία και πάλι θα σας τα στείλω για τα έτη 2015 και 2016 και ελπίζω με τα τελευταία σημεία να κάλυψα σχεδόν όλες τις ερωτήσεις σας. Ευχαριστώ, λέει η Πρόεδρος. Παρακαλώ ε, αν έμειναν εκκρεμότητες να μας στείλετε γραπτό στις απαντήσεις σας. Ευχαριστώ πολύ ενδιαφέρουσες οι παρατηρήσεις και σίγουρα πολύ σημαντικό αυτό το στοιχείο ότι θέλετε να στυλβώσετε την εικόνα και να, να βελτιώσετε τη φήμη της τράπεζας. Και το τελικό λόγο θα έχει ο συγκεκριτής μας ο κύριος Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Αντιπρόεδρο του πια όλες τις απαντήσεις. Αν τυχόν ε, δεν έχουν καλυφθεί όλες οι ερωτήσεις, καλό τους συναδέλφους να τις υποβάλουν. Πάντα υπάρχει καλή διάθεση για συνεργασία και βεβαίως ε, κρατάμε και το ραντεβού ώστε να συμπεριλάβουμε και στη δική μας την έκθεση τις παρατηρήσεις μας που πιστεύουμε ότι θα επηρεάσουν ουσιαστικά τη δουλειά της ΕΤΕΠ και θα τη βελτιώσουν. Περιμένω περαιτέρω ανταλλαγή απόψεων και αρχίζουμε αμέσως στη δουλειά στη δική μας έκθεση. Σας ευχαριστώ πολύ. 1η Φεβρουαρίου προβλέπεται να συστήσουμε την έκθεση του αδέλφου βάλει 6 Φεβρουαρίου για τις ε, τροπολογίες και στη, στα τέλη Φεβρουαρίου για την Επιτροπή. Για δε την Ολομέλεια προβλέπεται να εξεταστεί και να ψηφιστεί τον Απρίλιο προς το παρόν. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώσαμε την ημερήσια διάταξη. Ευχαριστούμε που είσαστε εδώ για την εντατική ανταλλαγή απόψεων. Στα διάφορα δεν βλέπω να έχει δίσει κανείς το λόγο. Σας καλώ την προσεχή Δευτέρα στις 3 η ώρα στη συνεδρίαση της Επιτροπής μας με αλλαγή στην ημερήσια διάταξη και κλεισμένο των θηρών θα συνομιλήσουμε την ΕΑΖΟ και βέβαια υπάρχει και ε, συνεδρίαση σύντον στον ε, Καλή επάνωδο και το ξαναλέμε την επόμενη εβδομάδα.